και μπορεί να μας μιλήσει για το θέμα του. Έχει έρθει ο κύριος Άρνολτ. Είναι παρόν ο κύριος Τόμ Άρνολτ, ο πρόεδρος ειδικής ομάδας για την αγροτική Αφρική. Θα καταφτάσει ανα πάσα στιγμή. Θέλει να προσθέσει κάτι η αντιπρόεδρος της ΔΕΒΕ, μήπως όσο αναμένουμε τον κύριο Άρνολτ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Σικέρσκι. Είναι χαρά μου που είμαι εδώ. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας ε, ε, για την διοργάνωση αυτής της κοινή συνάντησης. Θα ακούσουμε και τον κύριο Άρνολντ, ο οποίος έρχεται ως ο Νούμπο για τις τελευταίες εξέλιξεις. Η πρόεδρός μας, Δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα για την ε, παρουσίαση του κυρίου Άρνολτ. Οπότε μου ζήτησε να την εκπροσωπήσω. Η δουλειά της ε, Task Force αυτής είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα για τη δική μας Επιτροπή και ε, είναι αποφασιστική σημασία ε, για την εταιρική μα σχέση με την Αφρική και κυρίω για την ανάγκη για επενδύσει στη δημιουργία θέσεων εργασία. Ήδη αυτή την εβδομάδα, τη Δευτέρα, στην Επιτροπή ε, Ανάπτυξη αποφασίσαμε κάτι τέτοιο. Τα καθήκοντα τα οποία έχει αναλάβει η Task Force και για τα οποία θα συμβουλεύσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πραγματικά ουσιώδου σημασία για την ανάπτυξη της Αφρικής. Εγώ καταρχάς θέλω να ακούσω τι θα μας πει ο κύριος Άρνολτ. Να δούμε τι ακριβώς συστήνει η Task Force. Αλλά να κάνω εγώ κάποια αρχικά σχόλια. Για τη δική μας την Επιτροπή όταν μιλούμε για την ε, ε, αγροτική Αφρική, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η επισητιστική ασφάλεια και η μείωση της φτώχειας. Αυτή είναι η βασική μας στόχη. Ο στόχος της ε, συνεργασίας μας με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Γεωργίας είναι να εξασφαλίσουμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί κατά τρόπον ώστε να μην πλήττει τις αναπτυσσόμενες χώρες και να μην τις εμποδίζει, να μην εμποδίζει την ανάπτυξη της τοπικής γεωργίας και των τοπικών αγορών, για παράδειγμα στην Αφρική. Πραγματικά Προσβλέπω στην ε, παρουσίασή σας για να μας πείτε ποιες είναι οι πτυχές που σας απασχολούν. Κυρίως για την ε, μείωση της φτώχειας, για την επιστηστική ασφάλεια, μια που αυτή είναι η βασική στόχη για την ε, πολιτική και για την ανάπτυξη στα πλαίσια της ΚΑΠ. για το 2018 είχαμε μια πράσινη επανάσταση στην ε, Αφρική που τονίζει την ε, ανάγκη για αλλαγή, για ανάπτυξη, ώστε να μειωθεί η φτώχεια και να εξασφαλιστεί η ε, επιστηστική ασφάλεια. Επίσης υπογραμμίζει ότι το εμπόριο και η εμπορική γεωργία μικρής κλίμακας είναι σημαντική για να αναπτυχθεί η, ε, για να υπάρξει ανάπτυξη στην Αφρική και να μειωθεί η φτώχεια. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη. Γιατί το μοντέλο για την επιτυχία δεν ε, βασίζεται στην ε, μόνο καλλιεργητική γεωργία ή στην γεωργία μεγάλης κλίμακος ή, για, ή στην καλλιέργεια μόνο για εξαγωγές. Να συνεχίσω. The African Union has defined some clear objectives. Αυτή η στόχη λοιπόν είναι ξεκάθαρη για την επιστηστική ασφάλεια, για την Αφρικανική Ήπειρο και υιοθετήθηκαν στην διακήρυξη του 2014. To end, hunger. Για να αντιμετωπιστεί η, η φτώχεια για να επιτύχουμε 6% ετήσια ανάπτυξη στον τομέα της γεωργίας για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για τουλάχιστον 30% των νέων και να υπάρξει τουλάχιστον 10% των δημοσίων δαπανών για την γεωργία. Δυστυχώς πολλές αφρικανικές χώρες δεν είναι καθόλου κοντά στο να φτάσουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Αξίζει λοιπόν να δούμε πιο στενά τις χώρες που έχουν κάνει μια αξιόλογη πρόοδο, όπως η Αιθιοπία, που έχει επιτύχει το στόχο του 6% για την ετήσια ανάπτυξη και όπου η, η φτώχεια μειώθηκε στο μισό. Αυτό τονίζει και τη σημασία του τομέα της α, ε, ε, γεωργίας και τη συμβολής του στη μείωση της φτώχειας. Είναι σαφές ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη ιδιωτική επένδυση, γιατί από αυτές μπορούν να εφεληθούν όλοι. Αλλά οι αναπτυξιακοί εταίροι και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα είναι ωφέλιμες για τις οικονομίες και για τους πολίτες της Αφρικής. Επίσης, είναι σαφές ότι η ανάπτυξη του αφρικανικού γεωργικού τομέα θα χρειαστεί και στεναρούς δημόσιους θεσμούς και δημόσιες επενδύσεις. Ο ιδιωτικός τομέας βεβαίως χρειάζεται, αλλά και ο δημόσιος τομέας χρειάζεται και η πολιτική βούληση χρειάζεται. Ας πούμε το παράδειγμα της Ασίας και της Ευρώπης, αυτό ακριβώς καταδεικνύουν. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις, ας πούμε πρόσβαση στην αγορά, απώλειες μετά την συγκομιδή και αποθήκευση και επεξεργασία επίσης που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Αφρικής. Άλλος ένα σημαντικός παράγοντας είναι η πρόσβαση σε πιστώσεις για εμπορικούς γεωργούς μικρής κλίμακας που δεν εξυπηρετούνται από τις εμπορικές τράπεζες και ούτε από ε, ιδρύματα, τραπεζικά ιδρύματα για μικροδάνεια έχει ξεκινήσει αυτό το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Επενδύσεων ε, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Βιώσιμης Ανάπτυξης και γι' αυτό θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε από τον κύριο Άρνολτ τι συστάσεις έχει να προτείνει η δική του Task Force ώστε αυτό το σχέδιο των επενδύσεων να είναι πιο επιτυχές για για τον τομέα της γεωργίας. Uh, finally, finally, I need to, to make uh, with... Επίσης, ένα σχόλιο που αφορά μόνο τα μέλη της Επιτροπής uh, Ανάπτυξης. Η προθεσμία για τις uh, τρεις ε, εκθέσεις για τον κανονισμό, για την ΚΑΠ τον οριζόντιο κανονισμό και τον τροποποιητικό έχει τροποποιηθεί, έχει παραταθεί και τώρα η προθεσμία είναι 12 Δεκεμβρίου. Ναι. Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Φερχάπερα. Όπως Αντιληφθήκατε, έχει έρθει ο καλεσμένος μας ο κύριος Τόμ ο πρόεδρος ειδική ομάδας για την Αγροτική Αφρική, που θα μας παρουσιάσει τα επιτεύγματα αυτής της ειδική ομάδας. Ε, έχουμε και τους εκπροσώπους της Επιτροπής του αλλά συμμετέχετε και σε άλλες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 έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω για την αγροτική Αφρική. Έχουν έρθει κάποιοι άλλοι συνάδελφοι από την Task Force Αγροτική Αφρική βρίσκονται στο βάθος της αίθουσας. Να σας πω που έχουμε φτάσει όσον αφορά την δουλειά μας. Ναι, θα πρέπει να σας τονίσω πρώτα-πρώτα ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το έργο μας, αλλά σύντομα οφείλουμε να το ολοκληρώσουμε. Οπότε να έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε να ακούμε απόψεις από το τι θα πρέπει να αποτυπώνει η έκθεση που θα συντάξουμε για το έργο μας. Και τώρα αυτά θέλω να σας εξηγήσω σε αυτή την κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών. Για δούμε πρώτα πρώτα αφορά το πολιτικό πλαίσιο που κινείται η Task Force μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η πολιτική δέσμευση της Ευρώπης προς την Αφρική έχει γνωρίσει ρυθμούς ε, που έχουν επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια για πολλούς λόγους και σε επίπεδο κρατικό και όχι μόνο. Και ο πρόεδρος ε, Γιούνκερ τότε που μίλησε για την κατάσταση ένωση το 2018 πρότεινε να υπάρχει μια συμμαχία των δύο επίρων ούτω ώστε να υπάρχει κάποιο είδου ε, συνεργασία, να υπάρχει κάποιο είδου ωφέλεια. our terms of... Οπότε το σημεία αναφοράς για το έργο μας ε, είναι αυτά τα οποία στα οποία αναφέρθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Μάιο αρχίσαμε τη διαδρομές και θα συνεχίσουμε και ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε σε εβδομάδες τον Δεκέμβριο. Όταν ανατενίζουμε το μέλλον της ε, Αγροτικής Αφρικής, τι βλέπουμε. Βλέπουμε αυτό που θα μπορούσε να είναι ένας ε, φακός διπλής εστίασης. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να δημιουργήσει η Αφρική θέσεις απασχόλησης για τον πληθυσμό της που συνεχώς αυξάνεται και τι μπορεί να γίνει όσον αφορά τα αγροδιατροφικά, τι μπορεί να γίνει στην Ήπεθρο, πώς μας συμβάλλουν αυτά στην επιτυχία των στόχων. Επίσης, Άλλο ερώτημα είναι πώς μπορεί η Ευρώπη να συμβάλλει σε αυτή την ε, συνεργασία με την Αφρική. Πάλι για την επίκριση αυτού του στόχου. Για να σας πω ποιο είναι, ποια, ποια είναι η τάξη μεγέθους. Πρόκειται για ένα πληθυσμό που συνεχώ μεγαλώνει και οι προβολές από τον ΟΗΕ λένε ότι θα πάει ο πληθυσμό από 1,2 δι το 2015 στο 1,7 δι το 2030 και στη συνέχεια το 2050 στα 2,5 δις, αλλά μεταξύ του 15 και του 50 η Αφρική θα έχει το 70% της συνολικής αύξησης του πληθυσμού της υδρογείου. Πολύ εντυπωσιακό αυτό. Αυτή η αύξηση του πληθυσμού οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για νέες θέσεις απασχόλησης και τώρα έχουμε κάθε χρόνο 20 εκατομμύρια που μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Το 2030 θα έχουμε πάει στα 30 εκατομμύρια άτομα ε, και 60% αυτής της ε, αύξησης του εργατικού δυναμικού αφορά την Ήπεθρο. Αυτά τα εντυπωσιακά στοιχεία μας οδήγησαν σε δύο συμπέρασματα. Πρώτα-πρώτα, ότι η βασική πρόκληση των ηγετών της Υπήρου τις επόμενες ε, δεκαετίες αλλά και χρόνια θα είναι το να μπορέσουν να δημιουργήσουν αρκετή απασχόληση για να απορροφήσει όλη αυτή την εργατική δύναμη και δεύτερον ότι στα αγροδιατροφικά και στα της υπαίθρου ε, θα πρέπει και εκεί να υπάρξει δημιουργία θέσεων απασχόληση. Οπότε αυτό που εξετάζουμε είναι τι πολιτικές χρειάζονται τόσο ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερες θέσεις απασχόληση. Είναι αλήθεια όμως ότι αυτοί οι τομείς κινούνται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μιας συγκυρίας πολιτικής και οικονομική που αυτή θα καθορίσει το τι θα γίνει. Οπότε, ευθύ εξ αρχή στην έκθεσή μα τονίσαμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε κάποιο είδου πρόοδο όσον αφορά τον έχει πολιτική, μακροοικονομική σταθερότητα, ήπειρο, να έχουμε καθαρή ενέργεια ε, στην Ήπειρο, να προστατεύσουμε τους φυσικούς πόρους της Ήπειρου και πιστεύουμε ότι οι ηγέτες στη συνεργασία με την Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα και έτσι θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να υπάρξει πρόοδος στα αγροδιατροφικά, τα γεωργικά, αλλά πρώτα πρώτα ας μην μπούμε τώρα στις λεπτομέρειες γιατί αυτό δεν είναι στην εντολή μας. Αυτό τώρα που θέλουμε να ε, προσέξουμε είναι τι γίνεται σε αυτούς τους τομείς που εξετάσουμε και να δούμε τι θα γίνει, τι μπορεί να γίνει, ούτως ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Αλλά για να το καταλάβουμε αυτό θα πρέπει να δούμε τέσσερα ζητήματα σημαντικά που θα πρέπει να αποτελέσουν πολιτικές ε, προτεραιότητες και προτεραιότητες στις πολιτικές μας. Εδαφική προσέγγιση, οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση, ε, να αναδείξουμε την ε, αλληλεπίδραση μεταξύ των αστικών και αγροτικών περιοχών. Έτσι, θα έχουμε θέσει απασχόλησης. Έτσι η ύπεθρος θα γίνει πιο ελκυστική για τον κόσμο που μείνει εκεί και δεύτερον. Προτείνουμε κάποια μέτρα τόσο ώστε να βοηθήσουμε τον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό στην ε, γεωργία της Αφρικής γιατί υπάρχει μεγάλη ποικιλία στην Αφρική από χώρα σε χώρα όσον αφορά την παραγωγότητα και την ανάπτυξη. Έχουμε κάποιε χώρε, με ψηλά επίπεδα ανάπτυξης που έχουν κάποιες ε, πολιτικές ε, μου δίνουν τον προϋπολογισμό έχουν θετικό περιβάλλον για γεωργούς και για την βιομηχανία. Ε, αυτό σημαίνει ότι ο σκοπός μας θα πρέπει να είναι να έχουμε πιο πολλές χώρες που να έχουν τέτοια υψηλά πρότυπα και επιδόσεις τρίτων. Συστήνουμε να υπάρξουν επενδύσεις και να αναπτυχθεί μια βιομηχανία παραγωγής ε, τροφίμων στην Αφρική που να είναι βιώσιμη και ακόμα αυτό δεν έχει γίνει. Τα πράγματα εκεί ε, δεν έχουν αναπτυχθεί ε, όσον αφορά τη μεταποίηση και άρα μπορεί η Αφρική να αναπτύξει τον ε, δυτικό τομέα, να γίνουν εκεί επενδύσεις, η βιομηχανία να ακολουθήσει μια λυσίδα αξίας, να βελτιωθούν τα πρότυπα για την των τροφίμων, να υπάρξει εμπόριο ενδοαφρικανικό και κατά τέταρτον. Διαπιστώνουμε ότι η προστασία των φυσικών πόρων και η διαχείριση αυτών είναι πάρα πολύ βασικά πράγματα για να υπάρχει μια βιώσιμη παραγωγή και να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Μπορεί να βοηθήσει η Ευρώπη όσον αφορά τη διαχείριση, όσον αφορά κάποιες ε, στρατηγικές ε, αντοχής ε, του κλίματος σε σχέση με τις πολιτικές για ανάπτυξη της υπαίθρου. Οπότε, θα επικεντρώνουμε σε αυτούς τους τέσσερις άξονες, σε αυτά τα τέσσερα θέματα, ώστε στο τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης μας, να διατυπώσουμε κάποιες προτάσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν από την Ευρώπη και την Αφρική σε συνεργασία και θα τονίσουμε ότι θα πρέπει να βοηθήσει η να βοηθήσουν οι νέοι και ο τομέας ο αγροδιατροφικός και επίσης οι δυναμικές περιοχές της υπαίθρου ε, επίσης θα έχουν κεντρικό ρόλο. Οπότε θα υπάρξει συνεργασία των δύο επίρων για βιώσιμες επενδύσεις και απασχόληση όπως πρότεινε ο πρόεδρος Γιούνκερ το 2018 και έτσι μπορούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης για αυτούς τους τομείς και αυτά θα καλυφθούν από την συμπαράταξη των επίρων και θα πρέπει, λέμε, σε τρία επίπεδα να λειτουργήσει αυτή η εταιρική σχέση. Μεταξύ των ε, ανθρώπων, μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή για τους γεωργούς, τους φορείς τους, τους συνεταιρισμούς τους και μεταξύ των κυβερνήσεων, οπότε θα πρέπει η εταιρική σχέση να οδηγήσει σε μια ευρεία ε, συνεργασία των κοινωνιών, των επιχειρήσεων, των κοινωνήσεων, να επιτύχουμε την ε, πρόοδο, η τεχνολογία να δώσει ευκαιρίες και επίσης εδώ έχει να διαδραματίσει ρόλο η πολιτική ηγεσία, η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε συνεργασία με τα κρατημέλη θα πρέπει να υπάρχει μια συνεκτική, συνεπής προσέγγιση και έτσι να έχουμε μια αυθεντική συνεργασία των δύο πύρων και έτσι να αντιμετωπίσουμε μία από τις πιο μεγάλες προκλήσεις του καιρού μας και το πιο σημαντικό κατακλείδι είναι ότι ελπίζουμε ότι η εστίαση του έργου μας όσον αφορά την ανάγκη για απασχόληση ε, στους νέους στην αγροτική Αφρική πρόκειται να αποτελέσει μια πολιτική προτεραιότητα γιατί το αξίζει. Και επίσης σας ευχαριστούμε που έτσι μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε για αυτό το θέμα γιατί και την ε, Δευτέρα το απόγευμα πήγαμε στο Συμβούλιο. Ήταν πολύ θετική ανταλλαγή απόψεων Οπότε και σήμερα αυτό το οποίο κάνουμε είναι συμπληρωματικό όσον αφορά αυτή μας την προσπάθεια και περιμένω να ακούσω τα δική σας συμβολή. Σας ευχαριστούμε. Παίρναμε στη συζήτηση. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, κυρία Χόιμπουχ. Ευχαριστώ, κύριε Άρνολτ, για την παρουσίασή σας. Χαίρομαι πολύ για την ύπαρξη αυτής της Task Force. Χαίρομαι που ε, και ο ε, Επίτροπος Χόγκαν ασχολείται με το θέμα αυτό, γιατί το θέμα της επιστημικής ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε καταρχάς την αντιμετώπιση της ε, πείνας που είναι πολύ σημαντική, κυρίως για την Αφρικανική Ήπειρο, αλλά και τις σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για, την, για το ότι θα υπάρχει στο μέλλον κυρίως πάρα πολύ περισσότερος πληθυσμός από ό,τι τώρα. Οπότε χρειαζόμαστε ε, οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να διαχειριστούν το μέλλον τους μόνοι τους. Ε, έχω κάποιες ερωτήσεις να κάνω. Καταρχάς, Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό για την παραγωγή τροφίμων στην Αφρική. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να δούμε τις μεθόδους για το πώς παράγονται τα τρόφιμα. Για τη ΦΑΟ υπάρχουν πρωτοβουλίες για το ε, scaling up και για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη συμμετοχή των πολιτών σε όλη αυτή τη δραστηριότητα αλλά και να τους ε, παράσχουμε οικονομική ασφάλεια. Ε, η γεωργία, η οικολογία πώς θα παρέμβει σε αυτό. Έχετε κάτι να πείτε, έχει κάποια βαρύτητα. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό σε αυτό το τομέα. Θα, βλέπ, θα δούμε βέβαια τι θα κάνει και η ΦΑΟ. Επίσης, το κλίμα ε, θα πρέπει μάλλον να ενσωματωθεί σε αυτή την έκθεση γιατί είναι ουσιώδους σημασίας κυρίως για την Αφρική και για μας βέβαια στην Ευρώπη αλλά για την Αφρική ιδιωτέρως και θα με ενδιαφέρε να μας ε, πείτε ε, πώς ε, θα γίνουν οι επενδύσεις και σε περιφερειακό επίπεδο ε, αν, υπάρχει, ε, αν, αν ε, συμπεριλαμβάνεται η επεξεργασία, τι γίνεται με τις πιστώσεις, την εκπαίδευση κτλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο, δυστυχώς θα σας κλείνω το μικρόφωνο όταν ξεπερνάτε το λεπτό. Κύριε Μαγκίνες. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ Τόμ για την παρουσίασή σου. Ε, ξέρω το βιογραφικό του και πραγματικά συμφωνώ με τα σχόλια του Πρόεδρου. Με την πείρα σου στη Γεωργία και τις γνώσεις σου, θέλω να σου υποβάλω δύο ερωτήσεις. Πώς έχει εξελιχθεί η κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύεις ότι η παρούσα της κατάσταση επηρέασε θετικά ή αρνητικά το δικό σου έργο στην Αφρική. Τι δάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από το παρελθόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την ανάπτυξη της γεωργίας και την αύξηση της παραγωγής των τροφίμων. Μπορείτε να διδαχθείτε από τα παραδείγματα αυτά και να βοηθείτε στο έργο σας στην Αφρική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το έργο για πολλούς και διάφορους λόγους αυτό που κάνετε στην Αφρική. Αν μη τι άλλο για ηθικούς λόγους. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την Αφρικανική Ήπειρο και Πραγματικά μα κόβει την ανάσα το μέγεθος του προβλήματος, μας προκαλεί πραγματικά δέος και χρειάζεται πραγματικά πολιτικό θάρρος από τα κράτη-μέλη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρουν τη σωστή απόφαση και να βοηθήσουν την ανάπτυξη στην Αφρική. Γιατί τα εγγόνια μας ε, θα υποφέρουν αν εμείς δεν λάβουμε τις σωστές αποφάσεις και δράσεις. Ο κύριος Άγνιο, ευχαριστώ. Κύριε Άρνουλ, θέσατε μερικέ ερωτήσει και θα αποπειρωθώ να δώσω κάποιες απαντήσει. Μα είπατε ποιο είναι το καλό μοντέλο, ε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εκεί. Πριν από 40 χρόνια είχα πάει εκεί, είχα ζήσει εκεί και πιστεύω ότι το μοντέλο των μεγάλων καλλιεργειών είναι καλό γιατί είχαμε ε, έναν αγροτικό κόμβο με 500 υπαλλήλους, ε, πολύ κοντά στην πρωτεύουσα. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι να, καταρχήν θα πρέπει να αποθαρρύνει τους Αφρικανούς γεωργού να χρησιμοποιούν γενετικώ τροποποιημένους οργανισμού και γονιδιακή διόρθωση, γιατί είναι πολύ θετικό. Αυτά, ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάνναγκαν. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε για την παρουσίαση και λυπάμαι που δεν είναι περισσότεροι συνάδελφοι να σας ακούσουν. Γιατί πολλοί στο Κοινοβούλιο παραπονιούνται για, τις, για τους μετανάστες που έρχονται στην Ευρώπη, όταν όμως συζητούμε για λύσεις για να βοηθήσουμε τον κόσμο να παραμείνει στις αιστείες του, ε, δεν έρχεται κανένας ε, να λάβει μέρος στη συζήτηση. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Ρωτήστε τι μπορούν να κάνουν οι ευρωβουλευτές, τι λύσεις μπορούν να προτείνουν. Κάτι που μονίμως ε, ανακύπτει και καταγόμενος από μια χώρα που έχει βιώσει λοιμό, ε, μπορώ να πω ότι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να συστήσει τον κόσμο. Δεν νομίζω, γιατί σε τελική ανάλυση ο καθένας θα πρέπει ε, να βρίσκει μόνος του την τροφή του και να αναπτύσσει τη γεωργία του από το να περιμένει να τον συστήσει κάποιος άλλος. Δεν είμαι χριστιανό από αυτήν την άποψη, αλλά καλύτερα αντί να δίνουμε τροφή σε κάποιον να τον διδάξουμε πώς θα βγάζει την, θα παράγει την τροφή του. Γιατί αν απλώς σητίζουμε κάποιον και σταματήσουμε την παροχή τροφής, τι θα γίνει. Θα χαθεί ο υπόλοιπος κόσμος. Ε, και το θέμα δεν είναι να ζητήσουμε τον κόσμο, είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο να ζητηστεί μόνο του. Αυτό καταφέραμε να το κάνουμε στην Ιρλανδία. Και δεν νομίζω ότι αντί να παράγουμε μόνοι μα τη τροφή μα, ήταν καλύτερο άμα περιμέναμε να ζητήσουν κάποιοι άλλοι. Η κυρία Νόιχλ. Ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ και θα μα απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ένα πράγμα με ενδιαφέρει εμένα. Όλοι σκεφτόμαστε πώ μπορεί να πάνε τα πράγματα καλύτερα στην Αφρική. Όποτε μιλώ εγώ με συναδέλφου, νομίζω ότι σκέφτονται ότι τα συστήματα, τα δικά μας, να τα εξάγουμε. Όπως κάνουμε εμείς δηλαδή την αγροτική πολιτική, να το κάνουν και στην Αφρική. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι η Αφρική χρειάζεται ένα τελείω διαφορετικό σύστημα. Το ίδιο γίνεται και με την ε, πώληση, ας πούμε, των ε, ε, σούπερ μάρκετ που δουλεύουν με πάρα, πολλούς, πάρα πολύ λίγους ανθρώπους εδώ. αυτή είναι, αυτά είναι ε, κομμένα και ρεμένα για τις δικές μας ανάγκες. Στην Αφρική θα πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερο προσωπικό σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Εσείς έχετε στο νου σας κάτι για ποιο είδους πολιτική γεωργική θα μπορούσε να λειτουργήσει στην Αφρική. Και δεύτερον, μιλούμε συνέχεια για τις εμπορικές συμφωνίες με την, με την Αφρική. Λέμε συνέχεια τι ωραία που φροντίζει η Ευρώπη, την Αφρική. Εσείς πώς βλέπετε την κατάσταση με τα e και υπάρχει δυνατότητα να διευρυνθεί η αφρικανική αγορά. Ουσιαστικά εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι καλό για την Αφρική, αλλά τελικά αυτό ίσως να μην είναι έτσι. Θα με ενδιαφέρει η απόψή σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντρία. Ευχαριστούμε κύριε Άννοντ για την ομιλία σας. Δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο σας. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Όπως είπατε, καταρχήν θα πρέπει να αποφύγετε τα λάθη που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας τα υπενθύμισε ο κύριος Άγνιου γιατί με την υπερβολική αύξηση της παραγωγικότητας Ουσιαστικά κόψαμε το σύνδεσμο μεταξύ γεωργίας, ε, διατροφής και ανθρώπινης υγείας. Δεν θα πρέπει και στην Αφρική να κάνετε τα ίδια λάθη που κάναμε στην Ευρώπη τα τελευταία 50 χρόνια. Επίσης, στην Αφρική έχουμε διαφορετικές ε, συνθήκε και διαφορετικέ καλλιέργειε. Και μεταφέροντας τι καλλιέργειες από την Ευρώπη στην Αφρική, μεταφέρουμε και τα προβλήματα. Και το θέμα της αγροτικής ε, ανάπτυξης περισσότερο ε, μας αναγκάζει να συμπαρασταθούμε στην Αφρική και να βοηθήσουμε να αναπτύξει τοπικές μεθόδους και όχι να εξάγουμε τις δικές μας, να εξάγουμε τις δικές μας μεθόδους. Και το θέμα είναι ίσως να περάσουμε από παραδοσιακά συστήματα, ε, προγράμματα ανάπτυξης σε προγράμματα διαπεριφερειακής εταιρικής σχέσης. Πιστεύετε ότι τέτοιου είδου εταιρικέ σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική θα είναι πιο υποφελεί από τι παραδοσιακέ αναπτυξιακέ συμφωνίε. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μίτση είναι επόμενο. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Με τον Τόμι και με την Task Force, με τους συνεργάτες του είμαστε σε στενή επαφή την κατάλληλη στιγμή ε, εργάζονται γιατί έδωσε το έναυσμα ο πρόεδρος Γιούγκερ για αυτήν την ε, εταιρική σχέση και θα έχουμε την συνάντηση της 18ης Δεκεμβρίου στην Βιέννη. Η σχετική έκθεση δεν αποσκοπεί στο να πει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο για να θρέψουμε τον κόσμο. Όχι. Θέλω να πει ότι θα πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι στην προσπάθεια για να βρεθούν ε, λύσεις σε κάθε χώρα, σε κάθε περιφέρεια. Επομένω υπάρχουν ελεκτικές ε, προτάσεις και ε, πολιτικές καινοτομία χρειάζεται, έχουμε και τεχνολογίες που θα πρέπει να προσαρμοστούν στα της Αφρικής και υπάρχει ε, αυτή η πυροτική προσέγγιση με, την, ε, ε, το χώρο ελευθερών εμπορίου. Έχουμε αντιλήσει κάποια μαθήματα. Πρόκειται για μια διαδικασία που είναι προσαρμοσμένη στην Αφρική, αλλά θα πρέπει βέβαια να υπάρξει εμπόριο μεταξύ των Αφρικανικών χωρών περισσότερο. Θα πρέπει να υπάρξει ολοκλήρωση στην Αφρική. Δεν θα πρέπει να υπάρχει προσέγγιση του κέντρου και των ακτίνων που ξεκινούν από το κέντρο προς τα έξω. Αντί 60-70% έχουν εμπόριο μεταξύ τους 15%. Εμεί τότε υπάρχει πρόβλημα εξάρτησης, μία αυτάρκειας, άρα θα πρέπει να έχει κανείς τοπικές, περιφερειακές αγορές. Ίσως θα πρέπει κανείς να ε, προβάλλει τα μοντέλα της ΚΑΠ. Μπορεί να βοηθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη όσον αφορά την εδαφική προσέγγιση. Τέτοια προσέγγιση θέλουμε οπότε θα ωφελήσουν οι προσεγγίσεις του τύπου του προγράμματος Leader για τις μικρότερες πόλεις και για την Ήπεθρο και έτσι να μην έχουμε αστιφιλία προς τις τεράστιες ε, πόλεις, προς τις παραγκουπόλεις γιατί εκεί οι νέοι δεν βρίσκουν ε, την απασχόληση που ονειρεύονται τώρα όσον αφορά τη βιώσιμη διατροφή τους. θα χρειάζεται πιο σφαιρική θεώρηση περισσότερη ποικιλία στη διατροφή. Κανείς δεν έφερε το θέμα της κακής διατροφής, του υποσυντισμού. Υπάρχει παγισαρκία, υπάρχει η διασπάθηση των τροφίμων. Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι νορολογική βόμβα μια επιρροπή που έχει τέτοιο δημογραφικό δίκτυο. Άρα χρειάζεται περισσότερη ποικιλία στη διατροφή. Αλλά και θα πρέπει όλα αυτά να είναι προσαρμοσμένα στο κλίμα. Τα περισσότερα προβλήματα της Αφρικής αφορούν τα δικαιώματα. Αναφέρθηκε αυτό στο υπαριθμό 9 θέμα μας. Ο κύριος Σάγκηνο τα είπε τα σχετικά με το έδαφος. Επίσης η πρόβαση, πρόσβαση στο νερό είναι θέμα κλειδί. Απλά κάτι να κάνουμε επίσης για την ε, ε, περίμωση των δασών. Είμαι βέβαιος ότι τις επόμενες εβδομάδες η Task Force και οι συνεργάτες της θα καταλήξουν σε κάποια μεστή έκθεση η οποία θα καταγράφει ποια είναι τα βασικά θέματα και επίση, τι θα πρέπει να κάνουν κάτι μέλη, συμβούλιο, κοινωνία, κοινοβούλιο, τι θα πρέπει να κάνουμε σε βαρική θεώρηση, ούτως ώστε να υπάρξει κάποια παρέμβαση βραχυπρόθεσμα, μέσο και μακροπρόθεσμα, σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση, αλλά και με τα κράτη της Αφρικής χωριστά. Να είμαστε οι πρωτοπόροι σε σχέση με την αλλαγή προτύπων που θα πρέπει να αγκαλιάσει η Αφρική. Τώρα, βραχυπρόθεσμα, εφόσον πάρα πολύ πρόθεσμα, έχουμε ένα σωρό ερωτήσεις και περιμένουμε τις απαντήσεις. Κύριε Άρνοντο, έχεις λόγο. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Λέναρτ Μίτσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις και να καλύψω μερικά κοινά σημεία σε μια ευρή απάντηση. Νομίζω ότι η λέξη κλειδί εδώ είναι η εταιρική σχέση. Νομίζω ότι αυτή είναι, αυτό είναι το θεμέλιο, το επίκεντρο της απάντησης. Όπως είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ στο μήνυμα για την κατάσταση της Ένωσης, αλλάζει το είδος της, η φύση της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Γιατί η σχέση μας προηγουμένως ήταν βοήθεια και εμπόριο. Τώρα έχει μεταλλαχθεί αυτή η σχέση και έχει αναβαθμιστεί η πολιτική της ποιότητα και αυτό θα πρέπει να είναι το σημείο αφετηρίας γιατί η Αφρική σε πολλούς τομείς έχει τις δικές της πολιτικές. Στην Γεωργία για παράδειγμα έχει δύο δεσμεύσεις, αναφέρθηκατε σε αυτό. Έχουμε τη διακήρυξη του Μανέμπο, αλλά και η διακήρυξη του 2013 Μαλέμπο διακήρυξη του Μαλέμπο του 2013. Οπότε έχει και η Αφρική αναλάβει δεσμεύσει και σε μεγάλο ή μικρό βαθμό τη στηρεί, αλλά θα πρέπει να τη στηρίσει καλύτερα και να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά θα πρέπει να έχει μια καλύτερη σχέση με την Ευρώπη και θα πρέπει να βοηθήσουμε την Αφρική να υλοποιήσει τους στόχους της, γιατί πρωταγωνιστής θα είναι η Αφρική, εμείς απλώς θα συμπαρασταθούμε στην Αφρική. Και μπορούμε να συμπαρασταθούμε και να βοηθήσουμε την Αφρική εν μέρη και χάρη στη δική μας πείρα. Η κυρία Μαγκίνες μίλησε για την κοινή γεωρική πολιτική και πώς αναπτύχθηκε την τελευταία 20 ετία και πώς εξελίχθηκε. Είναι αναφυσβήτητο ότι πριν από 20-30 χρόνια η κοινή γεωργική πολιτική ήταν επιβλαβής για τα συμφέροντα των Αφρικανών γεωργών, γιατί είχαμε τις εξαγωγικές επιστροφές, εξαγωγικές επιδοτήσεις και άλλα θέματα που ε, απέβαιναν εις βάρος των, Αφρικανών γεωργών. Τώρα αυτά αλλάζουν. Και αλλαγέ τα τελευταία 20 χρόνια διευκολύνουν αυτή την ε, μεγαλύτερη προσοχή που δίνουμε στην αγροτική ανάπτυξη, στο περιβάλλον, στην ποιότητα των τροφίμων και όλα αυτά είναι κάποια γενικά διδάγματα που μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και στην Αφρική προσαρμόζοντάς τα στις αφρικανικές περιστάσεις και συνθήκες. Οπότε αυτό είναι ένα τμήμα της απάντησης. Σε ό,τι αφορά ε, την αγροοικολογία, στη συνεργασία με τη ΦΑΟ και ούτω καθεξής, όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε επαρκώς υπόψη. Αύριο θα συναντηθώ με τη ΦΑΟ και ε, έχει κάνει πολύ καλό έργο και για τα θέματα της αγροοικολογίας αλλά και για τη μετανάστευση. Και αυτό επηρεάζει και το δικό μας έργο. Τώρα, στο θέμα της εταιρική σχέσης. Υπάρχει σημαντικό πολιτικό συμφέρον και της Ευρώπης να βοηθήσει την Αφρική να αναπτύξει τη δική της οικονομία. Αυτό είναι και συμφέρον της Ευρώπης. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι το κίνητρο της πολιτικής σας δέσμευσης. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και αν θα θρέψει τον κόσμο, δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής, να σητήσει να θρέψει τον κόσμο. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει το γεωργικό της μοντέλο και τη γεωργική της πολιτική και κυρίως την τελευταία δεκαετία έχει στραφεί σε μια πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων και της ε, διατροφής γιατί δεν έρχεται μόνο στην παραγωγή ε, επαρκών τροφίμων, αλλά και στην παραγωγή ασφαλών υγιεινών τροφίμων. Και αυτό είναι μια πολύ εύλογη ανησυχία και μπορούμε να την μπορεί να τη συμμεριστεί και η Αφρική. Σε ό,τι αφορά τα θέματα της γης, καταρχήν θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την πραγματικότητα ότι το μεγαλύτερο τμήμα της Αφρικανικής Γεωργίας ε, ε, είναι μικρές ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις όπου οι γυναίκες διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο και θα πρέπει να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα αυτών των μικρών εκμεταλλεύσεων και την ασφάλεια του γεωργικού του εισοδήματος. Τέτοιο ύφο θα θέλαμε στις συστάσεις μας. Αλλά δεν υπάρχουν εδώ ούτε απλές ούτε εύκολες απαντήσεις. Σίγουρα ε, θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα στις μικρές εκμεταλλεύσεις, θα πρέπει ταυτόχρονα να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, ώστε ο κόσμος και να μένει στη γεωργία, αλλά και να αυξάνει το εισόδημά του από άλλες δραστηριότητες. Αυτό συνέβη και στην Ευρώπη και θα συμβεί αναπόφευκτα και στην Αφρική. Και το θέμα της, βιομηχανικής, της αφρικανικής βιομηχανίας τροφίμων, που είναι υπανάπτυκτη αυτή τη στιγμή. Η ανάπτυξή της είναι πολύ σημαντική και, και έχουμε πολλά να πούμε, πιστεύω. Αλλά α, αυτό προποθέτει συμμετοχή όχι μόνο του ιδιωτικού, ιδιωτικού τομέα, αλλά και των κυβερνήσεων. Θα πρέπει οι κυβερνήσεις να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να προσελκύσουν τον ιδιωτικό κλάδο και να επενδύσει στην βιομηχανία παραγωγής τροφίμων. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα φυτογειονομικά, ασφάλεια τροφίμων για να είναι ευκολότερη εμπορία των αφρικανικών προϊόντων και φυσικά να ληφθεί υπόψη και λυσίδα αξίας ε, στο εμπόριο τροφίμων. Αυτά, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και σίγουρα μερικά ήταν πολύ εύστοχα και θα ληφθούν υπόψη στις περαιτέρω μας εκθέσεις και συστάσεις. Τα τελευταία μου σχόλια θα τα κάνω στα φιλανδικά. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Ευχαριστώ τους ε, συμμετέχοντες. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Άρνολντ. Ε, ό,τι καλύτερο εύχομαι στην δουλειά σας από εδώ και μπρος για να μπορέσουμε τελικώς να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και ευχαριστώ πολύ ε, για το γεγονός ότι μπορέσαμε σήμερα να συζητήσουμε αυτά τα θέματα από κοινού οι δύο επιτροπές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο και η παραγωγή τροφίμων είναι αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως για να μπορούν οι πολίτες να παράξουν ε, τρόφιμα από μόνοι τους. Ακούσαμε πολύ ωραία σχόλια και προτάσεις για το τι σημαίνει σε αυτή τη μικρή κλίμακα η γεωργία και όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ποιες είναι οι μέθοδοι παραγωγής. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τα δάση, τη φύση, τα εδάφη, δεν θέλουμε να μολύνουμε το έδαφος. Θα πρέπει πάντα να το αφήνουμε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι όταν το πήραμε για να ξεκινήσουμε την παραγωγή. Και βεβαίω πρέπει να σκεφτούμε και την εσωτερική αγορά και τη λειτουργία τη. Είναι σαφέ ότι πρέπει να μπορεί κανεί να ζει από την παραγωγή των ε, τροφίμων και να μπορεί να απολαμβάνει την παραγωγή του και του κόπου του. Ο κύριος Άρνολτ προς το τέλος έκανε μια πολύ ωραία περίληψη ότι χρειάζεται δηλαδή ευρεία συνεργασία και φυσικά Όντω έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι συμβαίνει στην ε, ε, αναπτυξιακή συνεργασία και στην παραγωγή. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για τη συζήτηση αυτή και νομίζω ότι μπορείτε τώρα να συνεχίσετε με την ε, δική σας συνεδρίαση. Αυτά από εμάς, Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε κυρία Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε την Επιτροπή ΔΕΒΕ, τη Γραμματεία και τη Επιτροπής ΔΕΒΕ για την προετοιμασία αυτής της κοινή συνεδρίασης των δύο επιτροπών και πάνω απ' όλα ευχαριστούμε τον κύριο Τόμ Άρνολτ. Και πραγματικά σας θαυμάζουμε περιόριστα για το έργο σας. και ελπίζω να έχουμε ακόμη μια φορά την ευκαιρία πριν τελειώσει η κοινοβουλευτική μας θητεία να σας καλέσουμε και να σας ακούσουμε στην Επιτροπή μας. Θερμά ευχαριστώ, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Και ολοκληρώνουμε εδώ την κοινή συνεδρία των Επιτροπών Άγκρη και Ντέβε και συνεχίζουμε... Συνεχίζουμε τη συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας γιατί μας έμεινε μια κρεμότητα από την ημερήσια διάταξη. Οπότε επανερχόμαστε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης Επιτροπής Γεωργίας. Σημείο 9. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Στέφαν Μπάκες και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, την κυρία Πούλκινεν. Καλώς ήρθατε. Το σημείο 9, επαναλαμβάνω, προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με την ευκαιρία της εβδομάδας για τα ανθρώπινα δικαιώματα την ε, δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αγροτών και άλλων ατόμων που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές και για τις παγκόσμιες προκλήσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη γεωργία. Όπως ξέρετε, συμμετέχουμε και εμείς ε, στην οργάνωση της ε, εβδομάδας για τα ανθρώπινα δικαιώματα επ' ευκαιρία της 70ης επαιτίου της διακήρυξης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό λοιπόν να λάβουμε και εμείς μέρος Επιτροπή Γεωργίας στα θέματα αυτά και γι' αυτό καλέσαμε τον κύριο Στέφανο Μπάξ που είναι ε, αρμόδιος ε, του προγράμματος για την λογοδοσία στη FIAN ε, International. ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα στη, στα τρόφιμα και στις, στα συναφή οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και έχουμε και την κυρία Πούλκιν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Καλώς ήρθε, κυρία Μπάξ, καλώς ήρθε, κυρία Πούλκινεν. Θα δώσω 10 λεπτά στον κύριο Μπάξ και 5 λεπτά στην κυρία Πούλκινεν. Ελπίζω να σας αρκούν. Λυπάμαι κυρία μου, εσείς έχετε λιγότερο χρόνο. Ο κύριος Μπάξ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μπορούσαμε να έχουμε απαντήσεις. Υπάρχει χρόνος. Α, ωραία, ευχαριστώ. Να απάντηση του Πρόεδρου. Thank you very much for, for inviting me on the committee. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση στη συνεδρίασή σας για να σας πούμε για τα της ε, ε, δήλωση των για τα δικαιώματα αυτών που εργάζονται στις ευρωπαϊκές περιοχές. Αυτά γίνανε στον ΟΗΕ, στην ΟΗΕ πριν από λίγες μέρες. Αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό σε λίγο. Πρόκειται για μία δήλωση. Η UNDRP αναφέρεται σε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντική για διάφορους λόγους. Για να δούμε πρώτα πρώτα κάποια στοιχεία, κάποια περιστατικά, πραγματικά. Και αφορά αυτούς που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές γενικά, αγρότες και άλλους αυτοί που φροντίζουν για την επιστημιστική επάρκεια και ασφάλεια για όλο τον κόσμο. Αυτοί μας σητίζουν. Μιλούμε για το 70% των διατροφών που αυτοί οι μικροκαλλιεργητές ε, παράγουν αυτό το 70% και φροντίζουν για την ποιότητα των ε, ειδών και επίσης έτσι προστατεύουν γενικώ τους φυσικούς πόρους. Και έτσι έμεσα αντιμετωπίζονται και η αλλαγή του κλίματος. Όπως ξέρετε, όλο ένα και περισσότερο εξαφανίζονται οι μικρές γεωργίες εκμεταλλεύσεις και στην Ευρώπη και παντού. Ακριβώς γιατί μεγαλώνουν ε, οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Έχουν πλέον εκτήματα που δεν έχουν μικρές, οπότε το εισόδημα όλα είναι και συρρυκνώνεται. Πολλές φορές είναι και κάτω από το όριο της φτώχειας, το κατόφλι της φτώχειας. Έχουμε επίσης συγκέντρωση της γης, υπέρ των μεγαλοκαλλιεργητών. Έχουμε την αρπαγή της γης παντού και γι' αυτό Υπάρχει προστασία ευξημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αλλού οι αγρότες και οι άλλοι που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν ε, άσκηση βίας, ε, τους διώχνουν από τη γη τους μέχρι και τους δολοφονούν. Και έχουμε ένα σώρο ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σκοτώνονται, προσπαθούν να προστατεύσουν τη γη αυτήν. Αυτά γίνονται παντού και στην Ευρώπη. Και σας παραπέμπω στο περσινό ψήφισμα με ευρεία πλειοψηφία. Είχε προβλήματα εδώ η δική σας επιτροπή. Αυτό για τη συγκέντρωση της γης. Όλα αυτά μας δείχνουν τις δυσμενείς διακρίσεις βάρος αυτών των αγροτών. Αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση η κοινή αγροτική πολιτική έχει συμβάλει. Στον σχηματισμό πολύ μεγάλων εκμεταλλεύσεων και στην εξαφάνιση των μικρών. Α, να σας πω και ένα άλλο ψήφισμα ένα άλλο το οποίο φέτος ε, ε, εγκρίθηκε όσον αφορά την παραβίαση των ε, γηγενών, αυτοχθόνων και την υφαρπαγή της γης. Αυτό αφορούσε και τη δήλωση για τα δικαιώματα. Οπότε κλείθη έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη-μέλη να προσχωρήσουν στην δήλωση του ΟΗΕ. Κάποια πιο συγκεκριμένα θέματα τώρα. Είπαμε τι γίνεται όσον αφορά τους Γεωργούς Παντού. Είπαμε ότι παράγουν μέχρι και 80% των ειδών διατροφής. Αυτοί οι χωρικοί, οι μικροί καλλιεργητές. Ταυτόχρονα όμως 80% του κόσμου πεινάει. Και αυτοί ζουν στην Ήπεθρο, σε γεωργικές περιοχές, αγροτικές περιοχές. Και αυτό είναι βέβαια ηρωνία. Στην υποσαχαρία Αφρική οι γυναίκες συμβάλλουν μέχρι το 80% ε, στην δουλειά που αφορά την ε, παραγωγή αυτών των ειδών διατροφής. Και στη Λατινική Αμερική μέχρι το 40% όσον αφορά την ε, προσφορά των διατροφής και παρά όλα αυτά τα σημαντικά στοιχεία οι γυναίκες δυσανάλογα υφίστανται τον υποσυντισμό, τη φτώχεια, την διατροφική ανασφάλεια. Μια που δεν έχουμε χρόνο, να μην σας πω τώρα τι γίνεται όσον αφορά την σχετική διαδικασία, Και θα σας πω απλώς τι γίνεται όσον αφορά την κρίση, τι έγινε με το 2007-2008, η Δία Καμπεσίνα που ήταν αυτό το κίνημα πρόθεσε την ε, δήλωση αυτή, την υπόθεση της δήλωσης ε, στο Συμβούλιο της Γενέβης, το, το Συμβούλιο του ΟΗΕ. Είχαμε τότε αυτή την ε, κρίση του 7 και του 8 που απετέλεσε αφορμή για συνειδητοποίηση του τι γίνεται και αφορμή για ανάληψη δράση. Να τώρα να μην δούμε τα ενδιάμεσα στάδια. Και πάμε σε αυτή τη διακυβερνητική ομάδα το 2012 και πάμε στο 2018. Και μόλις πριν δύο μέρες η τρίτη επιτροπή του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη που συζητά θέματα ανθρωπιστικά και κοινωνικά ενέκρινε αυτήν την δήλωση με αρκετά μεγάλη πλειοψηφία Πολλέ ήταν οι αποχές και επτά οι αρνητικές για τη δήλωση ψήφι το Δεκέμβρη θα γίνει η κύρωση αυτής στην Ολομέλεια βλέπετε τώρα ένα χάρτη, ο ο χάρτης είναι πιο εύρωτο από τα λόγια και βλέπετε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Αφρική και Ασία σχεδόν συνολικά, ολοκληρωτικά ήταν υπέρ αυτής της δήλωσης. Κάποιοι ξέρει στη Λατινική Αμερική, τρεις μεγάλες χώρες, Βραζιλία, Αργεντινή και Κολομβία απέσχον. Στη δε Ευρώπη, να, Πώς έχει η κατάσταση. Όπως είναι στο χάρτη του ΙΕ, αποτυπώνονται οι χώρες και όπως βλέπετε έχουμε πάρα πολλές ε, αποχές. Μόνο δύο χώρες ψήφισαν υπέρ της δήλωσης. Πορτογαλία και Λουξεμβούργο. Και τρεις ευρωπαϊκές χώρες ψήφισαν κατά. μόνο Βασίλειο, Σουηδία και Ουγγαρία. Ψήφισε υπέρ και η Ελβετία. Καλό σημάδι. Και άλλε χώρες, όπω το Μονακό, η Μολδαβία, η Λευκορωσία και η Σερβία ψήφισαν υπέρ. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι το ότι η δήλωση. Δεν αφορά μια εγωστική προσέγγιση για προστασία ε, συντεχνιακών συμφερόντων των αγροτών. Τ' άκουσα αυτό. Θα πρέπει κανείς να είναι πέρα αυτής της κίνησης γιατί αυτή η δήλωση αφορά όλους. Δεν είναι προστατευτισμός. Και σας εξήγησα γιατί εξαφανίζονται μικρές εκμεταλλεύσεις. Αυτή η δήλωση είναι κατά των δεσμενών διακρίσεων και είναι πάρα πολύ σημαντική για τη διατήρηση της βιοπικιλότητας στη Γεωργία. Προστατεύει επίση το έδαφος για να είναι υγιές. Βοηθάει στην απασχόληση στην ύπεθρο, την ανάπτυξη της Υπέθρου και κατακλή. Είδατε πως ψήφισαν τα διάφορα κράτη και έχω ένα μήνυμα προκλητικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είπαν ότι είναι πρωταθλητέ στα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι λένε. Όμως διαπιστώσαμε ότι η συντηρητική πλειοψηφία του δεν ψήφισαν ναι όπω ανεμένεται. Όμως τα πράγματα εξελίσσονται. Η Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αρχίσουν να συνειδητοποιούν ότι είναι αναγκαία αυτή η δήλωση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι που εξελίσσεται. Εχρειάζεται πάρα πολύ αυτή η δήλωση. Ευχαριστώ κυρία Πούλκιναν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ για να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για να εορτάσουμε την διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας ε, Εξωτερικών Δράσεων θα ήθελα να ξεκινήσω στηριζόμενη στο συμπέρασμα του συναδέλφου. Επιβεβαιώνω ότι όντως τα κράτη-μέλη είναι οι πρωτοπόροι στην, ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Κανένας δεν κάνει τίποτα περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι. Σε σχέση τώρα με αυτή τη συγκεκριμένη διακήρυξη και τα δικαιώματα των αγροτών και όσους ζουν στις ε, αγροτικές περιοχές, ε, κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερως, θεωρούμε πολύ σημαντικό, από την ευρωπαϊκή οπτική Μάλλον από αυτή την οπτική είναι που ξεκίνησε να εμπλέκεται ενεργά στι διαπραγματεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στι συζητήσει τη Ομάδα Εργασία για τα Δικαιώματα των Αγροτών και άλλων ανθρώπων που ζουν στις, ε, ε, στην Ήπεθρο για το σχέδιο αυτό τη δήλωση. Και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή είναι μια διακοινοβουλευτική ομάδα εργασία, άρα τα κράτη-μέλη είναι αυτά που την στελεχώνουν και βεβαίω εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση παίζουμε τον συντονιστικό ρόλο. Όπως αναφέρθηκε, η δήλωση αυτή ε, υιοθετήθηκε τη Δευτέρα. 119 μέλη το ΟΗΕ την υποστηρίξαν, αλλά πρέπει να πω ότι 49 κράτη-μέλη απέσχον λόγω συγκεκριμένων ανησυχιών που άπτονται της δήλωσης. Όντω η Ολυβία προεδρεύει και αναγνωρίζουμε ότι κάποιε από τι προτάσει που έχουμε υποβάλει έχουν ληφθεί υπόψη, έχουν υπάρξει κάποιε βελτιώσει στο κείμενο. Επίση, εκτιμούμε την ε, ε, επικοδομητική ε, προσέγγιση που έχει αναλυφθεί από, την, από το Συμβούλιο στη Γενέβη. Βεβαίω αυτό ε, ισχύει όχι μόνο για τα κράτη-μέλη τη Ένωση, αλλά και ε, για, την, ε, για μέλη του ΟΗΕ. Τώρα, για τα συλλογικά ανθρώπινα δικαιώματα που και το δικαίωμα να έχει κανείς γη, να καταχεί γη και αυτό πρέπει όντω να διευκρινιστεί στην δήλωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, ε, έχουμε ακούσει κάποιες ανησυχίες από τα κράτη-μέλη για κάποιες ασυνέπειες που υπάρχουν μεταξύ των ε, νομικών δεσμευτικών πολυμερών συμφωνιών και της δήλωση αυτής, κυρίως για τον τομέα του περιβάλλοντος. Παρόλο που αναγνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι νομικό δεσμευτικό μέσο, δεδομένης και της περιπλοκότητας αυτής τη δήλωση, θα προτιμούσαμε να ε, παρατεθεί η υιοθέτηση σε μια μεταγενέστερη συνεδρίαση της γενική συνέλευση. Ε, μια τέτοια παράταση θεωρούμε ότι θα μας δώσει περισσότερο χρόνο για να μελετήσουμε καλύτερα και να αντιμετωπίσουμε, να λύσουμε τα προβλήματα, αλλά δυστυχώς αυτή την επιλογή δεν την είχαμε. Ακόμη και αν ε, δεν μπορούσαμε να έχουμε πλήρη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δήλωση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επιμένει στη δέσμευσή τη να συνεργαστεί με όλου του εταίρου για να αντιμετωπίσει αυτά τα σημαντικά προβλήματα και την ανισότητα που υπάρχει και προσπαθεί να ε, εφαρμόσονται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, οικονομικά, κοινωνικά, όλων των ανθρώπων που ζουν στην ε, Ήπεθρο και σε αγροτικές περιοχές η ε, απόκτηση γη είναι πολύ σημαντικό ε, θέμα για τους ανθρώπους που ζουν στην Ήπεθρο, οπότε επιτρέψτε μου να σα πω τι κάνουμε εμείς ως προς αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμερίζεται την ε, άποψη ότι η άμεση πρόσβαση στην και η κατοχή της γης και τα προβλήματα που υπάρχουν οφείλονται στην ανεπάρκεια λογοδοσίας. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει συμμόρφωση στους κανόνε και στις ε, ε, οδηγίες και στις πολιτικές ε, σε διεθνές επίπεδο όπως αυτές για, για το θεματολόγιο του 2030 και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτού του θεματολογίου, τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε κάποιες προτάσεις για την ανάπτυξη που καθορίζουν τη στρατηγική για τα μελλοντικά χρόνια. Η πρόσβαση στην, στους πόρους και στην γη βεβαίως αποτελεί κομμάτι ομοφωνίας στη δήλωση. Επίσης, υποστηρίζουμε τις και κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη ε, κατοχή γης και τη χρήση των δασών και παρόλο που συνεχίζουμε να ζητούμε από τα κράτη να εφαρμόσουν τις αρχές αυτές, ε, ε, χρηματοδοτούμε προγράμματα αντίστοιχα με έναν ε, προπολογισμό 240 εκατομμύρια ευρώ. Όλες οι δράσεις ε, αναφέρονται στο φυλάδιο που δημοσιεύθηκε πρόσφατα ε, για την υπεύθυνη χρήση γης και για το πώς έχει κατάσταση για το 2019. Συμπερασματικά να σας πω ότι θα εφαρμοστεί μια πολυσχεδής προσέγγιση ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τη χάνουν σεβασμού και εφαρμόνονται και εφαρμόζονται και για τον τομέα της γεωργίας. Θα υποστηρίξουμε βεβαίω ε, ε, όσους υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς θα συνεχίσουμε να ε, δουλεύουμε πάνω στην ε, πίεση για την ε, παγκόσμια εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων. Βεβαίως προσβλέπω στα σχόλιά σα, Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό οι υπόλοιποι. Ε, κυρία Σένερα, ένα λεπτό, ούτε δευτερόλεπτο παραπάνω. Κυρία Σένερα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πραγματικά κρίμα, πολύ κρίμα. Μια φορά που επιτέλους μιλάμε για τα δικαιώματα των χωρικών, των αγροτών, των αγροτησών, ε, το κάνουμε σε πέντε λεπτά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για μια η νυφάλια συζήτηση. Πολλά δε που εμείς οργανώσαμε αυτή την εκδήλωση και αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Βία Καπεσίνα και τους εταίρους της για το έργο που έκαναν που κατέληξε σε αυτή την έγκριση της δήλωσης για τα δικαιώματα των αγροτών, των αγροτεσών και των εργαζομένων στην, στην Ήπεθρα ε, μιλήσαμε για την αρπαγή των γεών. Αυτό είναι μια πραγματικότητα δυστυχώς ακόμη και στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το φαινόμενο ε, βρίσκεται και στη δική μας Ήπειρο και όχι μόνο στις άλλες. Ε, επίσης, ε, ήταν συμφωνημένη η ψήφος και μάλιστα είχαμε μαζική αποχή των κρατών μελών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ψηφοφορία αυτής της δήλωσης. Μόνο η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο ψήφισαν υπέρ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτές τις δύο χώρες για την στρατευμένη θέση τους υπέρ της διακήρυξης για τα δικαιώματα των χωρικών και επίσης να πω ότι η δήλωση είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για να βάλουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των χωρικών, των αγροτών και αγροτησών ε, πάνω από τα ε, συμφέροντα του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και των πολυεθνικών που είναι υπεύθυνε για την αρπαγή των γεών ε, και την αρπαγή των φυσικών πόρων. Σας ευχαριστώ κύριε Χόιμπουχ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι όλη τη βδομάδα εδώ στο Κοινοβούλιο, την ημέρα που εορτάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν είναι κανένας εδώ στην συνεδρίαση. Βλέπετε πώς αλλάζουν τα όρια. Οι χώρες που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες και που πλήττονται περισσότερο συμφωνούν και εμείς βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Είναι πραγματικά δραματικό το μήνυμα που δίνουμε για ένα δισεκατομμύριο ε, ε, αγρότες αυτή την, ε, σε αυτόν τον κόσμο που πραγματικά την χάνουν διακριτικής μεταχείρισης και απειλούνται καθημερινά. Αναρωτιέμαι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν μιλούμε για τα δικαιώματα των αγροτών απέχει και δεν θέλει να συνδυάσει την ε, όλη διαδικασία μαζί με τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. Θα το ξαναπώ, ντρέπομαι. Πραγματικά τι βάρος έχουν οι μεγάλες πολυεθνικές απέναντι σε ένα δισεκατομμύριο ανθρώπινες ψυχές. Κυρία Μαγκίνες, ευχαριστώ και ευχαριστώ για την παρουσία σας. Λυπάμαι γιατί πρέπει να φύγω και έχουμε τριμερή διάλογο σε λίγο, θα κρατήσει τρεις ώρες. Είναι πραγματικά πολύ άτυχη στιγμή που οργανώσαμε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων και η μικρή προσέλευση επίση. δυστυχή. Ε, δεν θα σχολιάσω για την, την ψηφοφορία της δήλωσης γιατί δεν έχω αρκετές πληροφορίες αλλά Συζητήσαμε προηγουμένω με την ειδική ομάδα για την Αφρική και ίσω κάποιε ιδέε σα μπορεί να βοηθήσουν και αυτή την ειδική ομάδα. Και νομίζω ότι ίσω ήταν το πιο επικοδομητικό που θα μπορούσε να προκύψει από την απογευματινή συζήτηση στην Ιρλανδία. Μετά την απόκτηση ανεξαρτησία είχαμε μεγάλο πρόβλημα με την κατανομή των γεών και έχουμε ακόμη κάποιε εκκρεμεί ε, ε, αμφισβητήσει ε, και διεκδικήσει. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα τη γη και τη ιδιοκτησία γη και έχουμε σε πολλές περιοχές ε, εμπόλεμες καταστάσεις, κανένα δικαίωμα του λαού στη γη και πραγματικά γι' αυτά θα μπορούσαμε να συζητάμε πολύ περισσότερο και να εντρυφήσουμε. Κύριο κύριος ευχαριστώ. Πολύ γρήγορα. Λυπάμαι από αυτές οι δύο συζητήσεις και για την πείνα στον κόσμο αλλά και για τα δικαιώματα των αγροτών. Ακολούθησαν ε, την συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ε, Είχαμε πολύ πιο εκτενή συζήτηση προηγουμένω και μας έμεινε ελάχιστος χρόνος για αυτές τις πολύ σημαντικές συζητήσεις. Γιατί ως προς τη διάγνωση των απειλών συμφωνούμε, ως προς μεθόδους τους διαφωνούμε. Επίσης, ε, μιλήσαμε για το θέμα της επιστηστικής ασφάλειας και της επιστηστικής κυριαρχίας. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων και είναι προαπαιτούμενο Έχουμε τα στοιχεία και τους λόγους ε, για τους οποίους η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απήχαν ε, και δεν υποστήριξαν τη δήλωση αυτή για τα δικαιώματα των αγροτών. Ε, αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει και στο μέλλον, γιατί το 2050 θα έχουμε 1 δισεκατομμύρια κατοίκους στον κόσμο. Πώς θα τους θρέψουμε. Οπότε δεν θα πρέπει αυτή η αύξηση της παραγωγής να, ε, που θα απαιτηθεί να γίνει βάρος των Ευρωπαίων γεωργών. Και σίγουρα η οικογενειακή γεωργία θα είναι μία από τις λύσεις ε, που θα πρέπει να διερευνήσουμε και στη συνέχεια των συζητήσεων στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία πολύ σύντομη απάντηση με τρία στοιχεία για να απαντήσω και στις απορίες των Ευρωβουλευτών. Ε, μετά τα σχόλια και τις εκπροσώπου της Ε.Ε. Τα επιχειρήματα των ευρωπαϊκών χωρών για να μην ψηφίσουν υπέρ ε, και να κρατήσουν τάση αποχή στη δήλωση για τα δικαιώματα των αγροτών ήταν τριπλά. Καταρχήν δεν θέλουμε συλλογικά δικαιώματα και